η οροθετική ασθενή τους. Και η κοινωνία θα ε, πρέπει να μπορεί να προστατεύεται, όχι μόνο οι άρρωστοι. Ευχαριστώ κύριε Κλάις Με την παρέμβαση αυτή ολοκληρώνεται ε, ο γύρος των επεξηγήσεων ψήφου. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους όσοι ε, έλαβαν το λόγο. και που τηρήσατε και τους χρόνους. Γι' αυτό δεν χρειάστηκε ουσιαστικά να διακόψω κανέναν παρεμβαίνοντας. Έχω λάβει από το Συμβούλιο δύο κοινέ θέσεις για πρώτη ανάγνωση, ε, καθώς και τους λόγους που τις οδήγησαν να το εγκρίνουν μαζί με τις αντίστοιχες θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τίτλοι θα ανακοινωθούν στα πρακτικά της παρούσης συνόδου και η τρίμηνη προθεσμία που διαθέτει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αποφανθεί αρχίζει από αύριο 2011. Τα πρακτικά της εχθεσινής και σημερινής συνεδρίασης θα υποβληθούν στο Κοινοβούλιο προς έγκριση στο Στρασβούργο και αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις ε, θα διαβεβασω στα όργανα που είναι αποδέκτες τα όσα αποφασίσαμε σήμερα με αυτή την παρατήρηση κηρύσω ε, τη διακοπή της περίοδου συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της πέρας συνεδρίας. Ευχαριστώ πολύ.